Και ήθελα να επισημάνω ότι ε, δεν είναι μια μεμονωμένη κίνηση αυτή, αλλά αντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια. Απευθυνόμενη στα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. Η 0065 του 2010 που υποβλήθηκε από τους συναδέλφους Βιντάλ, Κουάντρας, Σόντεργαν, Σίβενσον και άλλους για το Κάμπα Ραφ και, αυτό, και αυτή έχει πλειοψηφία από τον αριθμό των μελών του Κοινοβουλίου και γι' αυτό βάσει του άρθρου 123 του κανονισμού θα αποσταλεί στους ε, παραλήπτες. Ζητά το λόγο ο κύριος Στίβενσον, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές ε, που υπέγραψαν ε, την δήλωση 75 για το στρατόπεδο Άσραφ που αποστέλει ένα σαφέστατο και ισχυρό, ισχυρό μήνυμα στις αρχές του Ιράκ έτσι ώστε να τερματίσουν ε, την πολιορκία την παράνομη πολιορκία που έχουν αναπτύξει βάρος 3.400 ανθρώπων που βρίσκονται πολιορκημένοι μέσα στο στρατόπεδο Ασράφ. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που μας ε, υποστήριξαν σε αυτή τη συλλογή υπογραφών που ξεκίνησε μόλις πριν από ένα μήνα και που ε, σημείωσε τεράστια επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Στίβενσον. Να περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες. Ε, Προπολογισμό για το 2011. Τροπολογία υπαριθμών 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ.